κληρονομιά του Ευρωπαϊκού Έτους Ανάπτυξης. Εξ ονόματος του Συμβουλίου, το λόγο έχει ο κύριος Σμιτ. Παρακαλώ κύριε Σμιτ, έχετε το λόγο. <laughs> Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές, λίγες μέρες πριν τερματιστεί το έτος για την ανάπτυξη. Ε, χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί σας. Έχουμε ένα παράδειγμα εξαιρετικής συνεργασίας ανάμεσα στα ευρωπαϊκά όργανα, τα κράτη-μέλη, την κοινωνία των πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα και όλους όσους ε, L'Union européenne se sont très είναι κάτι το οποίο ε, θα έλεγα συγκεντρώνει το έτος για την ανάπτυξη όλους αυτούς τους πρωταγωνιστές. Νομίζω λοιπόν ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έχουν ε, μπορέσει ήδη από τον Ιανουάριο του 2015 να προχωρήσουμε λοιπόν στις οργανώσεις αυτές στα πλαίσια μιας κοινή προσπάθειας για την κοινή αξιοπρέπεια ε, και την κοινή πρόοδο, δρώντας μαζί με τα κράτη-μέλη σαν ε, παγκόσμιος εταίρος και φυσικά και σαν πρωτοπόροι στον τομέα της δημόσιας αναπτυξιακής βοήθειας και στα πλαίσια της συζήτησης που έγινε στις Βρυξέλλες για την περίοδο μετά το 2015 την παρουσία και του Μπαν Πάρα πολλές χώρες μέλη οργάνωσαν μεμονωμένα ένα, τα επίσημα εγγένεια θα έλεγα αυτής της νέας προσπάθειας για το 2015 ανανεώνοντας τα μέσα που διαθέτουν για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου πολλές χώρες έπαιξαν κομβικό ρόλο ε, φέρνοντας τις δραστηριότητες αυτές όσο πιο ε, κοντά γίνεται στους πολίτες. Συνεργαζόμαστε λοιπόν με τους τοπικούς εταίρους, με την κοινωνία των πολιτών, με όλους αυτούς τους εταίρους με τους οποίους έχουμε κοινές ευθύνες και κοινή αίσθηση αλληλεγγύης και φυσικά και τον ιδιωτικό τομέα. Ο ρόλος του είναι ως και η ευθύνη ανήκει σε όλους. Ε, δώσαμε ε, ιδιαίτερο βάρος στα κοινωνικά μέσα και γενικά στην ψηφιακή κάλυψη των ε, συγκεκριμένων αυτών οργανώσεων ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για τους νέους. Πάρα πολλοί νέοι εμπλέκονται άμεσα στις προσπάθειες που γίνονται και πρέπει να τους στηρίζουμε και να τους ενημερώνουμε έτσι ώστε να προκαλούμε και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από πλευράς τους. Το 2015 θα έλεγα ήταν μια εμβληματική χρονιά ε, γεμάτη ε, διεθνή γεγονότα που συνδέονται άμεσα με την ανάπτυξη. Η Διεθνής Έκθεση στο Μιλάνο, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, η διάσκεψη για την χρηματοδότηση της ανάκτησης στην Άντισα Μπέμπα και το COP21 τώρα στο Παρίσι. Όλα αυτά είναι γεγονότα τα οποία μεγένθηναν ε, την προσπάθεια για το έτος αυτό και επέτρεψαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να γνωστοποιήσει με ακόμα μεγαλύτερη πειθό τις απόψεις της και τις δυνατότητές της. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω τις συζητήσεις που κάναμε μέχρι τώρα, ιδιαίτερα για τη μετανάστευση και την κρίση των προσφύγων. Η ανάπτυξη είναι πάντα το κλειδί και στην ουσία το άλλο πρόσωπο του νομίσματος, η άλλη πλευρά καλύτερα του νομίσματος της μετανάστευσης. Είχα τη δυνατότητα να το πω αυτό όταν συζητήσαμε για την αηφορία για την αηφόρο ανάπτυξη εδώ και λίγους μήνες, η καταπολέμηση της φτώχειας, η καταπολέμηση της απελπισίας που οδηγεί τους πολίτες να εγκαταλείψουν τις χώρες τους. Αυτή είναι η προτεραιότητά μας. Φέτος μπορέσαμε να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη στα πλεονεκτήματα της ανάπτυξης και συνεργασίας όχι μόνο για τους φτωχούς λαούς αλλά και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση παρά τους δύσκολους καιρούς τους οποίους περνάμε. Οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι υπέρ της ανάπτυξης για τη συνεργασία και νιώθουν αλληλέγγυοι με τους λιγότερο ευνοημένους λαούς. Το πνεύμα αυτό θα πρέπει να παραμείνει ζωντανό και η αίσθηση αυτή της αλληλεγγύης θα πρέπει να μεταφραστεί σε συγκεκριμένες πράξεις. Να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την κυρία Μακάβεν και τους συναδέλφους της από την Επιτροπή Ανάπτυξης που έκαναν πάρα πολλά για να πετύχει η ευρωπαϊκή αυτή χρονιά. Την επόμενη εβδομάδα θα συναντηθούμε στο Λουξεμβούργο για να κλείσουμε τη χρονιά αυτή. Να εκφράσω την ευαρέσκειά μου και για την διοργανική συνεργασία η οποία επέτρεψε μέσα σε λίγο χρόνο να υπάρξει μια κοινή δήλωση Συμβουλίου, Επιτροπής και Κοινοβουλίου που θα είναι η κληρονομιά αυτής της χρονιάς για την ανάπτυξη. Η δήλωση αυτή επίσημα και συμβολικά θα υπογραφεί την 9η Δεκεμβρίου στο Λουξεμβούργο και έτσι θα μείνει αν θέλετε ένα γραπτό από την φετινή προσπάθεια που θα πείσει τα κράτη-μέλη να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους και πέραν της 31ης Δεκεμβρίου. της Επιτροπής, το λόγο έχει ο κύριος Μίμητσα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, προσεγγίζουμε το τέλος του Ευρωπαϊκού Έτους Αναπτύξεως, που υπήρξε ένα έτος εταιρικής προσπάθειας διαδικτύωσης μοιράσματος των εμπειριών. Είδαμε να συνέρχονται οι ευρωπαϊκοί θεσμοί με εθνικές κυβερνήσεις, με την κοινωνία των πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα, διεθνείς οργανώσεις, για να σπρώξουν το μήνυμα ότι η συνεργασία είναι αναγκαία και προς το συμφέρον όλους, όλων. Συγγνώμη. Το μέλλον μας εξαρτάται από αυτό και μας θυμίζει ότι η συνεργασία για την ανάπτυξη δεν ωφελεί μόνο τους ανθρώπους της αναπτυσσόμενης χώρες. Είναι και το πώς ανταποκρίνονται οι Ευρωπαίοι στις ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Επιθυμώ να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο για τον κρίσιμο ρόλο που έπαιξε στην ανάληψη πρωτοβουλίας και στην στήριξη και στην πρόθεση του Ευρωπαϊκού Έτους Αναπτύξεως. Αυτό έλαβε πολλές μορφές. Είδα και την πλατεία που έχετε πίσω από το κτίριό σας να είναι στολισμένη με αφήσει. Ευχαριστώ ιδίως τον πρόεδρο Μάρτιν Σούλτς τον πρόεδρο, την πρόεδρο μάλλον της Επιτροπής Αναπτύξεως κυρία και τον αντιπρόεδρο κύριο Σαλ Γκέρενς για την ισχυρή υποστήριξη που έδωσαν. Το 2015 υπήρξε κρίσιμο έτος για την ανάπτυξη με την ατζέντα δράσης της Άντις και την ατζέντα για την ε, βιώσιμη ανάπτυξη που εγκρίθηκαν καθώς ελπίζω επίσης ότι θα εγκριθεί και ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των αλλαγών του κλίματος. Ταυτόχρονα η αντιμετώπιση των ισχυρών ρευμάτων μεταναστών και προσφύγων μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να αντιμετωπιστούν οι ρίζες της αστάθειας και της παράτυπης μετανάστευσης. Με άλλους λόγους να δώσουμε στον κάθε ένα και στην κάθε μία τη δυνατότητα να ζήσει στην πατρίδα του ή στην πατρίδα της με αξιοπρέπεια και όχι να αναγκάζεται να διαφύγει απέναντι σε απάνθρωπες συνθήκες. Για μένα η επιτυχία του έτους αναπτύξεως ήταν και είναι η συνεταιρική σχέση με τόσους πολλούς φορείς και στην Ευρώπη και εκτός αυτής. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισαν όλοι μαζί την κληρονομιά του έτους αυτού στηρίζοντας μια κοινή δήλωση στην επίσημη τελετή λήξη στο Λουξεμβούργο. Α συνεργαστούμε, α συνεχίσουμε τη συνεργασία για να διατηρήσουμε αυτό το πνεύμα της εταιρική σχέση της συνεργασία και πέρα από την 31η Δωδεκάτου του τρέχοντο. Ας πάρουμε την κληρονομιά της Ευρωπαϊκή Χρονιά ανάπτυξη και α την προχωρήσουμε να γίνει το κοινό πλαίσιο, η πλατφόρμα για μια συνεχιζόμενη προσπάθεια ευρωπαϊκού διαλόγου για την ανάπτυξη και για τα επόμενα χρόνια. Περνούμε στον κύκλο των ομιλητών εκ μέρου των πολιτικών ομάδων. Για την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος το λόγο έχει για δύο λεπτά ο κύριος Στίερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, στις αρχές ε, το 2015 ελπίζαμε ότι θα ε, άλλαζαν τα πράγματα το 2015 και κάποιοι ίσως ισχυριστούν ότι χαρακτηρίζεται το έτος από τη μαζική μετανάστευση. Για άλλους είναι το έτος της ανάπτυξης. Σίγουρα είναι επικρατούσα τάση μεταναστευτική, αλλά όσα συνέβησαν επιβεβαιώνουν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε αποτελεσματικές αναπτυξιακές πολιτικές Πρέπει να εστιαστούμε στις ρίζες του προβλήματος ε, της μαζικής μετανάστευσης και συγκεκριμένα στη φτώχεια. Ε, αυτό μας οδηγεί σε συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε φαινόμενα διαφθοράς στις γειτονικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιήσαμε το Ευρωπαϊκό έτος Ανάπτυξης για να επιλέξουμε τους 16 στόχους που θα θέσουμε για να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά και τις ε, ρίζες ε, του προβλήματος ε, της μετανάστευσης. Το σημαντικό μετά τη σχεδίαση των στόχων είναι η υλοποίηση του θεματολογίου. Για την περίοδο μέχρι το 2030 θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στον αναπτυξιακό στόχο υπαριθμών 16. Σίγουρα θα πρέπει να βασιζόμαστε σε μια αναπτυξιακή πολιτική που περιστρέφεται γύρω από το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν θα υπάρξει ανάπτυξη χωρίς ειρήνη και τα Χρειαζόμαστε την ειρήνη και την ασφάλεια ταυτόχρονα. Θα ήθελα να συγχαρώ και τους συναδέλφους από τις υπόλοιπε πολιτικές ομάδες που συνεργάστηκαν στην Επιτροπή Ανάπτυξης και τον κύριο Γκέρενς που δραστηριοποιήθηκε ιδιαίτερα για την πρόθεση του ε, έτους ανάπτυξης. Ε, κάρτα τον κύριο Τσάνη. Τη Παρακαλώ κύριε Τσάνη, έχετε 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ για την ε, ευκαιρία που μου δίνετε να σας υποβάλω ένα ερώτημα. Δεν θα ήθελα να αμφισβητήσω αυτά που είπε ο συνάδελφος ότι άλλαξαν τα δεδομένα το 2015. Λέτε ότι χωρίς ειρήνη δεν μπορεί να νοηθεί ανάπτυξη. Μάλιστα. Όμως είδαμε ότι χωρίς ανάπτυξη, αντίστροφο, ότι χωρίς ανάπτυξη δεν υπάρχει ειρήνη. Η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα τώρα να ακολουθήσει μια εξωτερική πολιτική που βασίζεται στην ανάπτυξη. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως μόλις είπα, δεν νοείται ειρήνη χωρίς ανάπτυξη και το αντίστροφο. Αυτό είπα. Είναι, συμβαδίζουν τα δύο και υπάρχει ε, μια άρεκτη σχέση ανάμεσα στην ανάπτυξη και την ειρήνη αλλά και την ασφάλεια. Έχουμε λοιπόν ένα νέο θεματολόγιο τώρα αναπτυξιακό μέχρι το 2030 και αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να ε, διαπιστώσουμε στα πλαίσια της αναπτυξιακής μα πολιτικής ποια μέτρα πρέπει να μεταρρυθμίσουμε, πώς μπορούμε να άρουμε τους φράγμους για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και να προωθήσουμε και την ασφάλεια και την... Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η κυρία Μακάβαν για ένα λεπτό. Um, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω ένα λεπτό σήμερα. Γι' αυτό δύο σύντομα μηνύματα. Το πρώτο, δράση. Εμείς ξεκινήσαμε λέγοντας ότι πρέπει να κάνουμε πράξεις και να μην μείνουμε στα λόγια. Το κάναμε. Πήγαμε στην Άντις, πήγαμε στο Παρίσι. Ελπίζουμε λοιπόν να υπάρξει συμφωνία στο Παρίσι τις επόμενες μέρες στα πλαίσια του νέου προγράμματος δράσης. Αυτές όμως ε, οι υποσχέσεις πρέπει να γίνουν πραγματικότητα. Πρέπει να υπάρξει μια ουσιαστική κληρονομιά της προσπάθειας που κάναμε φέτος, όπως είπε και ο Επίτροπος και ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια νέα σχέση ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους για τα επόμενα 15 χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και την Λουξεμβουργιανή Προεδρία, τη, Λου... Προεδρία, τον Επίτροπο Μίμητσα, και όλους τους συναδέλφους που στήριξαν την προσπάθεια. Των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Σούλικ. Σας ευχαριστώ. Το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης είναι το αποτέλεσμα καλού μάρκετινγκ. Δύο τρίτα του πληθυσμού στην Ευρώπη θεωρούν ότι πρέπει να αυξηθούν οι δαπάνε για την αναπτυξιακή βοήθεια παρά την παγώδη αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δαπανά τόσα χρήματα για το μάρκετινγκ για να προωθεί τον εαυτό της ε, ε, περισσότερα από ότι η Coca-Cola σε παγκόσμια κλίμακα και τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν μεγάλα κομμάτια του ΑΕΠ τους. Η Φιλανδία φτάνει και το 0,6%, η Γαλλία το ίδιο. Ε, δεν είναι ρεαλιστικό να ζητάει κάποιος από χώρες όπως η Γαλλία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα που έχουν υψηλότατα δημόσια χρέη να ε, δίνουν 0,7% του ΑΕΠ για αναπτυξιακή βοήθεια. Ας σταματήσουμε να ονειρευόμαστε και να θεωρούμε ότι η Ευρώπη θα σώσει τον υπόλοιπο κόσμο. Ας είμαστε ρεαλιστές. Μία μπλε κάρτα από την κυρία Χαούταλα. Τη δέχεστε. Παρακαλώ, έχετε 30 δεύτερα κυρία Χαούταλα. Θέλω να ρωτήσω τον συνάδελφο αν ξέρει ότι οι συνάδελφοί του από το ε, αδελφό κόμμα στην ε, Φινλανδική Βουλή υποστήριξαν αυτή την πρόταση για το 0,7% του ΑΕΠ. Εσείς συμφωνείτε. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί διαφωνείτε. Έχετε 30 δευτερόλεπτα κύριε Σούλικ να απαντήσετε. Άνω, σάμας στην Βεβαίως, Και η Φινλανδία πλήττεται από ύφεση και πρέπει να παλέψει για να αντιμετωπίσει τα δικά της προβλήματα και όντως θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί. Το, αυτό που πρέπει να αποφύγουμε είναι να μεγαλώσει το δημόσιο έλλειμμα. Μόνο με χρηστή ε, δημοσιοοικονομική διαχείριση μπορούμε να ε, προσπαθήσουμε να ε, λειτουργούμε ως ήρωες και να σώζουμε τον υπόλοιπο κόσμο. Κρατών, το λόγο έχει για δύο λεπτά ο κύριος Γκέρενς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μετά από 11 μήνες εκστρατείας και ευαισθητοποίησης μπορούμε να πούμε ότι το Ευρωπαϊκό Έξι ήταν επιτυχές. Υπήρξε συνεργασία ανάμεσα στους βασικούς πολιτικούς εταίρους στους εκπροσώπους των μη κυβερνητικών οργανώσεων και του ιδιωτικού τομέα. Οι μεγάλες προκλήσεις τις οποίες είδαμε το 2015 απέδειξαν την συνεισφορά της ανάπτυξης στην επίλυση πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, όπως το προσφυγικό. Πρέπει λοιπόν η αρχή του σεβασμού της αξιοπρέπειας ε, να είναι και ήταν στο κέντρο της εκστρατείας 2015. Κάποιες χώρες μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σεβάστηκαν αυτή την αρχή. Άλλες προώθησαν την αρχή της αδιαφορίας. Κανένα όριο, καμία ποσόστοση, καμία προσπάθεια να γίνει σεβαστή η αξιοπρέπεια. Έτσι λοιπόν τα προβλήματα της ανισότητας, της κακής διακυβέρνησης, της απειλής της εσωτερικής ειρήνης στις υποανάπτυξη χώρες είναι αποτέλεσμα και αυτών που κάναμε εμείς τα τελευταία 15-20 χρόνια. Είναι το αποτέλεσμα της δράσης μας και κυρίως της μη δράσης μας. Ας ε, μην αγνοήσουμε λοιπόν τις εξελίξεις τις οποίες μπορούμε να επηρεάσουμε για τα επόμενα 20 χρόνια. Ας είμαστε αποφασιστικοί. Έχουμε δώσει την υπόσχεσή μας. Η υπόσχεση θα πρέπει να την σεβαστούμε δεν θα πρέπει να τερματίσουμε την τεράστια προσπάθεια ευαισθητοποίησης του 2015. Ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας. Θα συνεχίσουμε και μετά το 2015. Ας δράσουμε λοιπόν σύμφωνα με τους στόχους αυτούς, τις αρχές αυτές, η κοινή δήλωση του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής είναι ένα θετικό βήμα. Για την ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, το λόγο έχει για 1,5 λεπτό η κυρία Σάντσες Καρντελντέι. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Δεν θα ήθελα να πω ότι ήταν θετική, να κάνω ένα απολογισμό θετικό ή αρνητικό. Πάντως ήταν το 2015 ένα πολύ σημαντικό ε, έτος Υπήρξαν πολλές συναντήσεις ε, ε, σε σχέση με την επίτευξη των στόχων που έχουν θέσει τα Ηνωμένα Έθνη και την επόμενη εβδομάδα ελπίζουμε να υπάρξει ένα φιλόδοξο σχέδιο για την καταπολέμηση ε, των κλιματολογικών συνεπειών. Η προσπάθεια την οποία κάνουμε είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ελπίζω το 2015 να μην μείνει ένα κενό να υπάρξει συγκεκριμένη δράση. Οι στόχοι μέχρι το 2030 έχουν καθολικό χαρακτήρα, θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να κάνουμε πραγματικότητα τα μέτρα. Θα πρέπει να ε, φροντίσουμε τις πολιτικές αυτές, τις πολιτικές για την ανάπτυξη και τότε δεν θα πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά που κάνουμε τώρα, να δίνουμε με το ένα χέρι και να παίρνουμε με το άλλο ε, φτωχαίνοντας τους λαούς του Νότου. Θα πρέπει ε, να πετύχουμε τους στόχους τους οποίους έχουμε μέχρι το 2030 και τότε το 2015 μπορεί να θεωρηθεί σαν μια ουσιαστική αλλαγή. Τον λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα που εγγράφηκε στην ημερήσια διάταξη είναι ασφαλώς πολύ σημαντικό. Στην Γερμανία έχω συμμετάσχει σε πολλές εκδηλώσεις όπου συζητήθηκε το εμπόριο, η μετανάστευση, κυριαρχία και τα όσα γίνονται και όσα δεν γίνονται. Είναι επίσης σημαντικό να καταδείξουμε και τα όσα έχουμε ήδη αναλάβει και επιτελέσει εδώ, χωρίς ωστόσο να μπορούμε να επαναπαυθούμε, διότι τα λόγια τώρα πρέπει να τα ακολουθήσουν οι πραγματικές πράξεις για να εξασφαλιστούν τα δικαιώματα των ανθρώπων και ιδίως το μέλλον των παιδιών μας. Εδώ πρέπει να δράσουν οι εθνικές κυβερνήσεις βεβαίως, αλλά και ο κάθε πολίτης. Σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, ασφαλώς πρέπει να γίνει σεβαστή η αξιοπρέπεια των ανθρώπων αυτών. Πρέπει να είναι καλόδεκτοι στις χώρες μας και πρέπει να είμαστε πρόθυμες και πρόθυμοι να αναζητήσουμε κοινέ λύσεις. Σε ό,τι αφορά το SDG, πρέπει να αρχίσουμε εμεί οι ίδιοι πρώτα-πρώτα να μειώσουμε την κατανάλωσή μας, να μειώσουμε τα απορρίμματα και δεν χρειάζεται ειδικό τίτλος του Πρωθυπουργού. Ο κόσμος μας ο ίδιος σημαίνει για να διατηρηθεί πρέπει να ξεπεράσουμε εαυτούς, πρέπει να αγνοήσουμε τα ίδια τα δικά μας τα συμφέροντα. Συνοχή της πολιτικής. Στην ομάδα Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας το λόγο έχει ένα λεπτό ο κύριος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να εκφραστώ θετικά όπως ε, μίλησαν αρκετοί συνάδελφοι γιατί είναι αλήθεια ότι κατά κάποιο τρόπο χρησιμοποιήσαμε τους πόρους που έχουμε για να κάνουμε διαφήμιση περισσότερο και όχι για να μιλήσουμε για την πραγματική ανάπτυξη. Παρόλη την κρίση για τους πρόσφυγες, ε, παρόλη την αύξηση των μεταναστευτικών ροών, στην ουσία απαιτείται πολύ περισσότερη δύναμη και μέσα για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα για την ανάπτυξη εκτός Ευρώπης. Παρ' όλα αυτά λοιπόν κάποια πετύχαμε, δείξαμε ότι μέχρι τώρα δεν υπήρξε ουσιαστική εφαρμογή των αρχών και των προγραμμάτων που έχουμε μέχρι σήμερα αποδεχθεί. Ελπίζουμε στο μέλλον να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα Τώρα δεν είναι βέβαια η στιγμή για να κρίνουμε τα αποτελέσματα, αλλά περισσότερο για να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Όπως ε, είπε και η κυρία Καλτεντέη, ε, στην ουσία η εμπορική πολιτική είναι αυτή η οποία καθορίζει το πώς θα υπάρξει πολιτική ανάπτυξη. Ομιλητών εκ μέρους των πολιτικών ομάδων για την ομάδα των Εθνών και της Ελευθερίας το λόγο έχει για 1,5 λεπτό ο κύριος Στούγκερ. Ευχαριστώ κύριε, Πρόεδρε. Πρόεδρε. Βεβαίως, τότε η χρονιά δεν είναι η μόνη χρονιά για την ανάπτυξη. Από τότε που άρχισε να λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει πολλά χρήματα για την ανάπτυξη. Ποια είναι όμως τα αποτελέσματα. Τα χρήματα πηγαίνουν για παράδειγμα στους δικτάτορες της Ζιμπάμπουε, της Μοζαμβίκης και της Σιέρα Λεόνε. Όλα τα λεφτά που πήγαν στον Μουγκάμπε τι έκανε, μπάρμπεκιου έκανε με κρέας ελέφαντα. Δύο ελέφαντες. Πρέπει να αρχίσουμε να κοιτούμε πραγματικά που πηγαίνουν τα χρήματά μας. Χρήματα πολλά πήγαν στη Ζιμπάμπου, επιμένω, και τα κράτησε για τον εαυτό του. Ο πρόεδρος Γκαμπών αγόρασε ακίνητα στο Παρίσι με τα χρήματα αυτά. Υπάρχει λοιπόν μια σχέση εξάρτησης ανάμεσα σε κυβερνήσεις και πολίτες. Βεβαίως η κυβερνήσεις χρειάζονται φόρους, του οποίου πληρώνουν οι πολίτες. Οι πολίτες όμως δεν θέλουν να καταβάλουν φόρους σε ανεύθυνες κυβερνήσεις. Αν λοιπόν η κυβέρνηση είναι διεφθαρμένη και λαμβάνει βοήθεια από την αλλοδαπή, όπως αυτές οι κυβερνήσεις που προανέφερα, μπορεί να συνεχίσει να κυβερνά χωρίς να εισπράττει φόρους. Επομένως εκεί τα πράγματα αυτά πάνε χέρι με χέρι και έτσι στηρίζονται οι διεφθαρμένοι δικτάτορες. Αυτά πρέπει να αλλάξουν. Θα έπρεπε να λέγεται έτος της διαφθοράς. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εδώ στις Βρυξέλλες ε, εξετάζουμε την έκθεση και ψηφίζουμε τον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης και ένα χρόνο μετά γίνεται μια συζήτηση και ένας απολογισμός για το πρώτο έτος ανάπτυξης. Είχαμε τη δυνατότητα για ένα ολόκληρο χρόνο να ενημερώσουμε τους συμπολίτε μας για τα τις 12 θεματικές ενότητες ε, προτεραιότητας, να τους εξηγήσουμε με ποιο τρόπο χρησιμοποιούμε τα χρήματα των φορολογουμένων, με ποιο τρόπο μέσα από το ε, Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης μπορούμε να αλλάξουμε την καθημερινή ζωή των ε, πολιτών, των φτωχότερων κόσμων ε, συγγνώμη, φτωχότερων κρατών της Ευρώπης και του κόσμου. Η Ρουμανία λοιπόν είναι από τις φτωχότερες χώρες της Ευρώπης. Εκεί όμως δυσκολευτήκαμε να δούμε τη σύνδεση ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης και τη βελτίωση της ε, καθημερινής ζωής ε, των πολιτών. Ε, είμαι συνεισηγητής και ήθελα να τονίσω, μιλώντας για αυτό το πρώτο Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης, ε, πρέπει να γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια για να εξηγήσουμε στους συμπολίτε μας περί τίνος πρόκειται. Πρέπει να επενδύσουμε στο μέλλον μας. Ε, δεν είναι θέμα επικοινωνιακής πολιτικής είναι ουσιαστικό το ζήτημα για να υλοποιηθεί το θεματολόγιο 2030 χρειάζεται άμεση εμπλοχή πολλών φορέων, άμεση συμμετοχή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εάν δεν δράσουν, δεν θα μπορέσει να σημειωθεί πρόοδος. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Γκερέρο Σαλόμου. Ε, Ευχαριστώ πολύ. <clears throat> Απαιτείται να υπάρχει λίγο μεγαλύτερη συνεκτικότητα και στα πλαίσια του διοργανικού διαλόγου και καλύτερη συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους ε, ε, κράτησε συγκεκριμένες ε, θέσεις. Προσπαθήσαμε. Παρ' όλα αυτά το Δεκέμβριο έχουμε περισσότερα προβλήματα από ό,τι τον Ιανουάριο. Περισσότερες κρίσεις, περισσότερες συγκρούσεις και απαιτείται να υπάρξει απάντηση πιο φιλόδοξη από ό,τι προηγουμένως. Το θέμα δεν είναι να είμαστε γενναιόδοροι απλά. Θα πρέπει να υπάρξει η όθηση έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις με αποφασιστικότητα. Θα πρέπει καταρχάς να ολοκληρώσουμε την προσπάθειά μας έτσι ώστε να φτάσουμε στο 0,7% του πλούτου μας για να βοηθήσουμε αυτούς οι οποίοι ζουν ουσιαστικά στο 0,7% της δικής μας ευμάρειας. Λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Σουζαντόφσκι. E, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υποστηρίζω σε μεγάλο βαθμό την αναπτυξιακή βοήθεια. Όπως ο Πάπας Παύλος δεύτερος ανανέφερε, είναι βασικός ρόλος αυτός της Ευρώπης να βοηθά τις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Όμως δεν θα πρέπει να είναι θέμα μάρκετινγκ και επικοινωνιακής πολιτικής. Ε, πρέπει συγκεκριμένα να αποτιμήσουμε τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού ε, Έτους Ανάπτυξης και να αναρωτηθούμε οι δαπάνες μας στην αναπτυξιακή βοήθεια αντιστοιχούν στις ανάγκες ε, των αναπτυσσομένων χωρών. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι μεγάλοι φορείς ε, στη διεθνή κοινότητα ε, όπως η Κίνα και η ΙΠΑ που συνδυάζουν τις προσπάθειές τους ή θα έπρεπε να συνδυάζουν τις προσπάθειές τους με τις δικές μας. Δεν είναι θέμα image, είναι θέμα συγκεκριμένων αποτελεσμάτων και αλληλεγγύης. Ε, θα έπρεπε να τροποποιήσουμε και την εξωτερική μας πολιτική για να αποκριθούμε στις προκλήσεις. Ευχαριστώ. Θα ακολουθήσει η κυρία Άντερσεν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος δωρητής βοήθειας στον κόσμο. Αλλά από τα χρήματα αυτά πόσα πάνε στην ανάπτυξη, πόσα χρήματα ανταυτού πηγαίνουν σε στρατιωτικές δαπάνες και σε πολέμους. Ευρωπαϊκό έτος ανάπτυξης βοήθησε στο ξερίζωμα της φτώχειας. Αντίθετα, τα μέτρα αυτά συμβάλλουν στην ανάπτυξη της, στην αύξηση της φτώχειας με ε, χρηματοδότηση πολέμων. Ρίχνουν ακόμα περισσότερες βόμβες στη Συρία. Δεν είναι ούτε απάντηση ούτε λύση αυτό το πράγμα. Αυτά οδηγούν σε περισσότερους θανάτους, περισσότερους ε, πρόσφυγες. Τέτοιοι πόλεμοι δεν αφήνουν παρά ερήπια. Χιλιάδες παιδιά χωρίς σχολεία, αθώα θύματα και πολλά λεφτά στις τσέπες των εμπόρων όπλων. Χρειαζόμαστε στόχους ανάπτυξης που να αναγνωρίσουν ότι η φτώχεια δεν είναι καμιά φυσική θεομηνία, ότι υπάρχουν λόγοι και αίτια για αυτήν. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος Βίλαντ, ευχαριστώ κύριε Άντερσεν, η Χαουταλά. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Καθώς λύγει το έτος της ανάπτυξης σιγά σιγά, αρχίζουν φιλόδοξες διαπραγματεύσεις για συμφωνία για το κλίμα. Θα ήθελα να εφιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι χρειάζεται να επενδύσουμε περισσότερα στην προσαρμογή όλων στις ε, αλλά που προκαλεί η αλλαγή του κλίματος, ιδίως για τις χώρες της Αφρικανικής Σαχέλ που είναι εντελώς απροστάτευτες όταν ε, επέρχονται οι αλλαγές του κλίματος πιστεύω ότι πολλές από τις δυνάμεις της αγοράς δραστηριοποιούνται για ένα μετριασμό των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος. Δεν οδηγούμαστε όμως σε πραγματική προσαρμογή. Αυτό είναι ένα κενό. Ευχαριστώ κυρία Χαουταλά. Επιτρέπετε να σας θέσει ο κύριος Στούγκερ ερώτηση. Δέχεστε την ερώτηση του κύριου Στούγκερ. Ορίστε κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ερώτηση. Μιλούμε εδώ και για ε, πρόσφυγες και για κλίμα. Τα αναμειγνύουμε όλα αυτά. Χειροτερεύει το κλίμα, γι' αυτό χρειαζόμαστε έξτρα αναπτυξιακή βοήθεια και παρόλα αυτά έρχονται οι πρόσφυγες. Όλα αυτά βέβαια συνδέονται. Η αλλαγή του κλίματος, εγώ είμαι Ολλανδός, ως χώρα είμαστε πολύ ευέλικτοι. Εμείς στην ουσία είμαστε κάτω από το επίπεδο της θάλασσας. Μήπως πρέπει να μας δώσετε κάποια από τα λεφτά μας πίσω από όλα αυτά που έχουμε δώσει για αυτό το τσίρκο. Ευχαριστώ η κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ ε, για την δήλωση που κάνατε. Εγώ πιστεύω ότι οι κάτω χώρες είναι σε θέση να βοηθήσουν τις πραγματικά φτωχές χώρες του κόσμου να προσαρμοστούν στην αλλαγή του κλίματος, διότι εσείς διαθέτετε τις κατάλληλες τεχνολογίες. Και αυτό που αναμένει ο κόσμος από μας στη διαπραγματεύση για το κλίμα είναι οι πλούσιες χώρες να διαθέσουν τις τεχνολογικές εξελίξεις που διαθέτουν, δηλαδή που έχουν δηλαδή στα χέρια τους, όχι μόνο για τον έλεγχο των πλημμυρών, αλλά και επενδύσεις σε ανανεώσιμες ενέργειες και στην αποδοτικότητα της ενέργειας. Αυτά είναι πράγματα που οι Ολλανδοί τα γνωρίζετε πολύ καλά και μπορείτε να βοηθήσετε με τον τρόπο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χαουταλά. Α, ναι, ναι. Ε, ε, δεν έβρισκα το κουμπί για να σας διακόψω. Όταν επιτρέπω γαλάζιες κάρτες να αναμένετε ότι στα 30 δευτερόλεπτα θα σας διακόπτω, χωρίς κτυπήματα του σφυριού κτλ. Εσείς κύριε Γκίλ τώρα. Ένα λεπτό. Δεν έχετε μικρόφωνο κύριε. Αρχίστε από την αρχή. Φέτος, το 2015 δηλαδή, υπήρξε το Ευρωπαϊκό Έτος της Ανάπτυξης. Είμαι βέβαιος ότι όσοι μας παρακολουθούν στο YouTube και εκείνοι τρεις απάνω εκεί στα θεωρία γνωρίζουν καλά τι σημαίνει αυτό. Αλλά ας γίνουμε ρεαλιστές. Όπως είχα προείπει πέρσι, αυτοί οι αυτοέπαινοι έχουν αγνοηθεί απολύτως από το κοινό στις χώρες μας τα 17 εκατομμύρια ευρώ που πετάχθηκαν από το παράθυρο θα μπορούσαν και θα έπρεπε να είχαν χρησιμοποιηθεί για να σώσουν ζωές όχι για να διαφημίσουμε πόσο σπουδαίοι και πόσο ε, καταπληκτικοί είμαστε με τα χρήματα των φορολογουμένων. Δεν θα υπάρξει καμιά κληρονομιά του Ευρωπαϊκού Έτους Ανάπτυξης. Ευχαριστώ κύριε Γκίλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης για μένα υπήρξε επιτυχημένο έτος γιατί έδειξε πόσο σημαντική είναι η πολιτική συνοχή για την πολιτική της ανάπτυξης. Αυτό κατέστη σαφές στους 12 ε, θεματικούς μήνες. Τα είδα αυτά και στη γερμανική Bundestag και ζήτησα να υπάρχει ε, έκθεση για τη συνοχή αυτή. Βεβαίως υπήρχαν και αρνητικές πλευρές στην Αντίσα Μπέμπα δεν καταφέραμε να επιτύχουμε το 0,7% από τις χώρες μέλη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να πανάτε δηλαδή για την αναπτυξιακή βοήθεια. Ταυτόχρονα και εδώ θα αντίπω στον συναδελφό μου, ήταν καλή η εκστρατεία γιατί έδειξε ότι στήσαμε στα πόδια της και μία ε, ε, συμμαχία για τα υφαντουργικά με συμμετοχή και του Συμβουλίου. Και αυτό αποτέλεσε και το προβάδισμα και για τους στόχους του 2020. Η συνοχή θα ενισχυθεί κι άλλο. Ευχαριστώ τον Επίτροπο αλλά και τους εκπροσώπους του Συμβουλίου για την πολύ επιτυχή εργασία και συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό, Σίλβα Περέιρα. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, επίτροπε, αυτό το ευρωπαϊκό έτος ανάπτυξης ε, δεν άλλαξε τον κόσμο, αληθεύει αυτό ε, και δεν το περίμενε και κανένας. Όμως άξιζε τον κόπο, ε, διότι υπήρξε ευαισθητοποίηση της κοινή νόμης, τροφοδοτήθηκε η συζήτηση και κυρίως προωθήθηκαν εταιρικές σχέσεις, προγράμματα και αποφάσεις που ακολουθούν τη σωστή κατεύθυνση. Όπως παραδείγματο χάρη σημαντικές διεθνείς διασκέψεις όπως εκείνη της Αντίσα Μπέμπα και της Νέας Υόρκης. Όμως τίποτα από αυτά που κάναμε δεν είναι χέγγιο για την επιτυχία. Η εφαρμογή των δεσμεύσεων στις αναπτυξιακές πολιτικές δεν είναι δεδομένη. Συχνά λείπει η πολιτική βούληση και υποστήριξη από το κοινό για την αναπτυξιακή πολιτική. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι ανησυχίας και πρέπει να είμαστε όλοι σε εγρήγορση να είμαστε σε γρήγορση και να απευθύνουμε μια έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς όλους τους ηθήνους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τόσο ώστε να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε Σίλβα Περέ. Περνάμε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye. Ε, δεν έχουμε χρόνο για όλους τους ομιλητές. Έχουμε διπλό αριθμό από αυτό για τον οποίο έχουμε χρόνο. Παρακαλώ, ε, δείξτε κατανόηση Ευχαριστώ. Κατά το Ευρωπαϊκό έτος ανάπτυξης νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι και κυρίως λαμβάνοντας υπόψη ε, τη μεταναστευτική κρίση και την COP21 συνειδητοποιήσαμε ότι είναι προς συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών να προωθήσουν την ανάπτυξη των φτωχότερων χωρών του κόσμου και να ε, ε, τόσο ώστε να αυξηθεί το επίπεδο ζωής ε, των πολιτών αυτών των χωρών, ε, ούτω ώστε να μην αποφασίζουν οι άνθρωποι να εγκαταλείψουν τη χώρα τους. Η μετανάστευση εξάλλου είναι επιζήμια πρώτα απ' όλα για εκείνες τις χώρες. Η μαζική μετανάστευση υπονομεύει τις αναπτυξιακές προοπτικές κάθε χώρας. Εκείνες οι χώρες θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια κυρίως σε εμπόλεμες ζώνες για να κρατήσουν κυρίως τους νέους ε, στη, στη χώρα ε, οι νέοι είναι αυτοί που ε, έχουν την ε, απαιτούμενη εκπαίδευση για να στηρίξουν τη χώρα και εκείνοι εγκαταλείπουν τη χώρα που δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα η αναπτυξιακή μας βοήθεια. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το 2015 έχει θεωρηθεί ως έτος υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάμεσα στους κύριους στόχους του Ευρωπαϊκού Έτου Ανάπτυξης είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων και της παραβίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η εμπέδωση του κράτου δικαίου και η οικοδόμηση δίκαιων και χωρί αποκλεισμού θεσμών. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να μην προωθεί την ανάπτυξη όσο θα έπρεπε στα κράτη-μέλη τη. Έτσι, για το 2015-2016 προβλέπονται 18,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε αναλήψει υποχρεώσεων, προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα για να έχουμε απασχόληση και ανάπτυξη. Το ποσό αυτό δεν είναι επαρκέ και θα πρέπει να αυξηθεί κυρίω για τι χώρε του Ευρωπαϊκού Νότου, που έχουν φτωχοποιηθεί από τη μερκελική λιτότητα όσο το χρέο ορισμένων κρατών μελών τη ένωση παραμένει στα τωρινά επίπεδα είναι αδύνατο να επιτευχθούν οι στόχοι του ευρωπαϊκού έτου ανάπτυξη. μόνο με τη διαγραφή του χρέου των χωρών αυτών και ιδίω με τη διαγραφή του επονίδιστου του χρέου στην ελλάδα θα μπορέσουμε να έχουμε ανάπτυξη να χτυπηθεί η φτώχεια και να τονωθεί η απασχόληση και η ευημερία. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Μαριά. Ο κύριος Γιάκοφτσιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. όλα τα τεκτενόμενα των κόσμων και όσα συνέβησαν το 2015 δείχνουν εν τέλει ότι το Ευρωπαϊκό Έτος Αναπτύξεως ήταν δικαιολογημένο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες μέλη της βοήθησαν όλες ε, τις χώρες και βοηθούν όλες τις χώρες που έχουν ανάγκη στον κόσμο. Η αλληλεγγύη, μάλλον δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή στην αλληλεγγύη. Υποστηρίξαμε εμείς το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης, όπως και υποστηρίζουμε και θα υποστηρίξουμε όλες τις προσπάθειες για να προληφθεί η μετανάστευση για λόγους κλίματος. Αυτή βεβαίω θα είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Ο κύριος Χρυσόγονος. Συζητούμε σήμερα για την αναπτυξιακή βοήθεια που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο λεγόμενο Τρίτο Κόσμο το 2015, στο πλαίσιο της οποίας υποτίθεται πως η θεματική έμφαση για το μήνα Δεκέμβριο θα ήταν στη σύνδεση ανάπτυξης και προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων όλα αυτά όμως ηχούν ηρωνικά όταν πριν από τρεις μόλις μέρες το ευρωπαϊκό συμβούλιο επιβράβευσε οικονομικά και πολιτικά το ημιαυταρχικό καθεστώς ερντογκάν στην τουρκία ξεχνώντας τις συστηματικές παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων. η στη μαζική δολοφονία εκατοντάδων ειρηνικών διαδηλωτών στην άγκυρα πριν μερικές εβδομάδες η δολοφονία του προέδρου του δικηγορικού συλλόγου του ντιγιάρμπακυρ πριν μερικές μέρες οι συλλήψεις δημοσιογράφων για αποκαλύψεις σχετικά με την υπόθαλψη των εγκληματιών του ισλαμικού κράτους από το καθεστώς ερντογάν όλα ξεχάστηκαν για την εξυπηρέτηση πρόσχερων σκοπιμοτήτων. το τουρκικό καθεστώς εμπορεύεται το προσφυγικό δράμα και η ευρωπαϊκή ένωση ακολουθεί πολιτική κατευνασμού εξευτελίζοντας το δικό της κώδικα αξιών. Ε, ε, ευχαριστώ κύριε Χρυσόγονε. Ο κύριος Έθριτζ. Thank you, Chairman. Um... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στο Ηνωμένο Βασιλείο η αναπτυξιακή βοήθεια είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενο ζήτημα. Ε, και παρότι γίνονται περικοπές στην άμυνα, στην παιδεία, στην επιβολή του νόμου, ε, στο σύστημα υγείας, ε, διαφυλάτουμε ακέραιη την αναπτυξιακή βοήθεια και όπως ε, έλεγε και ένας ε, πρώην ηγεμόνος μας, ε, δεν θα, θα θορυβηθούν οι πολίτες μας αν μάθουν ότι στέλνουμε τα χρήματα σε ένα μάτσο περίεργους δικτάτορες ανά τον κόσμο και ε, επίσης ότι θέλουμε λεφτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνέχεια μεταφέρονται αυτά τα χρήματα πάλι ε, σε αυτές τις χώρες. Ε, περισσότερα χρήματα δηλαδή των φορολογουμένων χρησιμοποιούνται και για την επικοινωνιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μας πούνε τι καλά ή που τα κάνουμε όλα που πράττουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Απαράδεκτο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κύριε Αθρέτζη. Ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πέρα από Ευρωβουλευτής είμαι και δήμαρχος σε μια πολύχνη της Βόρειας Ιταλίας και βλέποντας ε, τους ε, ισολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και τον προϋπολογισμό, κάθε φορά πρέπει να πάρω και ένα αλκασέλτσερ για να μπορέσω να δεχτώ και να χωνέψω αυτά που βλέπω. Στην Ευρώπη προσπαθούμε να προσέχουμε τις δαπάνες για να βοηθήσουμε τους πολίτες και όσους έχουν ανάγκη. Γι' αυτό είναι προσβολή να υπάρχουν τέτοιες δαπάνες. Δηλαδή στην ουσία μας χαρίζουν τα χρήματα δέκα δις ε, για την Τουρκία στην αρχή και τώρα δίνουμε κι άλλα. Όταν δούμε πώς λειτουργεί η Τουρκία είναι προσβολή να δίνουμε χρήματα. Και ξεχνάμε τους δικούς μας ανθρώπους στην Ευρώπη, τους Ευρωπαίους, αυτούς που καταβάλουν τους φόρους και θα πρέπει να λαμβάνουν πολλά χρήματα. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Εδώ λίγη η διαδικασία catch και στο τέλος των συζητήσεων λαμβάνει το λόγο πάλι ο Επίτροπος κ. Μίμητσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη. Στις αρχές του έτους γνωρίζαμε ότι το 2015 θα απέβαινε κρίσιμο για την χαρτογράφηση της μελλοντική ε, συνεργασίας για την ανάπτυξη η υιοθέτηση των νέων στόχων ανάπτυξης μας έδωσε το πλαίσιο για τις εργασίες μας για τα επόμενα 15 χρόνια. Ο κόσμος είναι όλο και πιο περίπλοκος και κινείται όλο και ταχύτερα. Νέες προκλήσεις εμφανίστηκαν φέτος για να μας θυμίσουν πόσο σημαντική είναι η ανάπτυξη και πώς πρέπει να λειτουργήσει αυτή ε, για την μετανάστευση. Η ανακοίνωσή μας για θέματα ανάπτυξης πρέπει να ανταποκρίνεται στην πρόκληση αυτή. Να συμμετέχουν σε αυτή όλοι οι ερκνό, ιδίω δε οι νέε και οι νέοι, για να στηρίξουν την ε, βιώσιμη ανάπτυξη και πέραν από το 2015. Ας χτίσουμε πάνω στα όσα πετύχαμε ήδη στο ευρωπαϊκό αυτό έτος για να εξασφαλίσουμε ώστε να συνεχίσει να ακούγεται η φωνή των πλέον ευάλωτων. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Τον λόγο στο όνομα του Συμβουλίου λαμβάνει ο Υπουργό κ. Σμιτ. Ευχαριστώ κυρίε και κύριοι. Επιθυμώ να ευχαριστήσω και πάλι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την συμβολή του στην επιτυχία του Ευρωπαϊκού Ετου Αναπτύξεω, που όντω λύγει τώρα. Ωστόσο οι προσπάθειε μας ε, για το ξερίζωμα τη φτώχεια θα πρέπει να συνεχιστούν και μάλιστα να ενταθούν Ιδίως πρέπει να μεταφραστούν πραγματικά μέσα από τη συνεργασία μας για ανάπτυξη σε, συγκεκριμένα, σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις οι οποίες οφείλουν να γίνουν σεβαστές. 1,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν ακόμα σε ακραία φτώχεια και ακόμα και αν εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι μπόρεσαν να βγουν από τον κύκλο της φτώχειας οφείλουμε να διαπιστώσουμε ακόμη ότι οι ανισότητες και μέσα στις ίδιες τις χώρες τους έχουν ε, γίνει ακόμα πιο σκληρές. Το ίδιο κινδυνεύει η επιβίωση του πλανήτη μας και από τις, αλλαγές, από τις επιπτώσεις της ε, αλλαγής του κλίματος. Πρέπει λοιπόν να γίνουν όλες οι δυνατές προσπάθειες τώρα στο Παρίσι ώστε να αντιμετωπιστεί η κλιματική πρόκληση. Διότι αυτή είναι και η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης. Άλλωστε δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς ανάπτυξη. Το είπατε και εσείς αυτό. Και δεν υπάρχει ασφάλεια σε έναν κόσμο όπου οι ανισότητες στην ανάπτυξη εξακολουθούν να παραμένουν τόσο σημαντικές. Θα πρέπει λοιπόν η δέσμευση αυτή υπέρ της ανάπτυξης να μην λήξει με την λήξη του έτους. Αυτή η προσπάθεια ευαισθητοποίησης και πειθούς πρέπει να συνεχιστεί με τρόπο ενεργό. Σας ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος Βίλαντ, σας ευχαριστώ. Κύριε Σμιτ, λίγη